τις γυναίκες εργαζόμενες. Ε, καλή εργασία εύχομαι σε όλους. Επίσης θέλω να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία βουλευτών της Ραλάνκα και της Μιανμάρ που είναι σε επίσκεψη εργασία στο Ευρωκοινοβούλιο για να μελετήσουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρίως του ελέγχου προπολογισμού. Siamo onorati Μας τιμά η παρουσία σας και σας ευχόμαστε καλή εργασία. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν από την ε, συνεδρίαση της 6ης Απριλίου